ίσο την επανάληψη της περίοδου της Συνόδου που διεκόπη στις 29 Μαρτίου. Αγαπητοί συνάδελφοι, χαίρομαι πάρα πολύ διότι σήμερα μπορούμε να καλωσορίσουμε για πρώτη φορά στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 12 Κροάτες παρατηρητές. Αξιότιμοι συνάδελφοι από την Κροατία, σήμερα για πρώτη φορά καταλαμβάνετε τα έδρανά σας στην αίθουσα αυτή της Ολομέλειας. Από αύριο θα συμμετέχετε στις συνεδριάσεις των Επιτροπών και των Πολιτικών Ομάδων συμμετέχοντας στις συζητήσεις. Έτσι την, ε, θα προετοιμάσετε καλά και θα παρακολουθήσετε την επικείμενη προσχώρηση της χώρας σας και θα μπορέσετε να εκπροσωπήσετε επάξια τα συμφέροντα της χώρας και των πολιτών της. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, όπως γνωρίζετε, ήδη επικύρωσε τη Συμφωνία ε, Ένταξης και ελπίζουμε ότι την 1η Ιουλίου του 2013 η Κροατία θα γίνει το 28ο μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα είναι ιστορική ημέρα αυτή για την Κροατία. Πιστεύω ότι θα είναι εξίσου ιστορική ημέρα για την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα Δυτικά Βαλκάνια γενικά. Κυρίες και κύριοι, Σήμερα συνεργάζονται ως παρατηρητές οι νέοι συνάδελφοι, αργότερα ως πλήρη μέλη. Αυτό σηματοδοτεί ότι παρά την κρίση που συζητούμε και πρέπει να συζητούμε καθημερινά, η Ευρωπαϊκή Ένωση ως ιδέα συνεργασίας κρατών και λαών πέραν των συνόρων δεν έχει χάσει την ελκτική της δύναμη. Εξακολουθούν να υπάρχουν πολλοί που ζηλεύουν αυτή τη διαδικασία ολοκλήρωσης. Υπάρχουν ε, κράτη και λαοί που θέλουν να ενταχθούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό πρέπει να το δούμε ως μεγάλη ευκαιρία και ως κατάφαση της ιδέας της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Γι' αυτό νομίζω ότι αυτό αποτελεί και ε, λόγο προβληματισμού σχετικά με το μέλλον της πορείας αυτής η προσπάθεια αυτή συμβολίζεται από τη σημερινή παρουσία των Κροατών παρατηρητών μας. Άλλη μια φορά ένα θερμό καλώς ήλθατε. Τα πρακτικά των συνεδριάσεων από 28 και 29 Μαρτίου και τα κείμενα που έχουν εγκριθεί υπάρχουν. Υπάρχουν αντιρρήσεις ως προς αυτά. Όχι, από ό,τι βλέπω, άρα λοιπόν τα πρακτικά εγκρίνονται. Ο κύριος Δήμητας Στογιάννοφ έκανε μια πρόταση από 8